Ε, εξέτασε τις εντολές των κυρίων Χοκ και Κλωσφόψκη και πρότεινε την επικύρωση των εντολών τους με ισχύ την 27η Νοεμβρίου 2015. Υπάρχουν ε,